So, es sind drei Kollegen anwesend, inklusive meiner Wenigkeit. Und ich würde vorschlagen, dass wir... Προτείνω λοιπόν να ξεκινήσουμε με το σημείο 18 της ημερήσιας διάταξης. Το θέμα εδώ πέρα είναι οικολογικού σχεδιασμός όσον αφορά τα συνδεδεμένα με την ενέργεια προϊόντα. Και έχουμε προσκαλέσει την Κομισιόν είχαμε θέσει μία ε, ερώτηση και θα δώσουμε τον λόγο στην Κομισιόν και μετά θα περάσουμε συζήτηση με τους ε, υπόλοιπους. Με τους δύο συναδέλφους. Ευχαριστώ. Είμαι, κάρ Κάρλο Πετινέλη και ασχολούμαι με την Γενική Διεύθυνση Επιχειρηματικότητας της Επιτροπής και μας ε, ε, ενδιαφέρει ολοκλήρωση και παρουσίαση της οδηγίας EcoDesign. Σα Σας ευχαριστώ γιατί μου δίνετε τη δυνατότητα να σας δώσω πληροφορίες για την αναθεώρηση της οδηγίας. Όπως γνωρίζετε, το Δεκέμβριο του 2012 η Επιτροπή ε, ενέκνε μία έκθεση ε, για την αναθεώρηση αυτής της οδηγίας, διά, δυνάμει του άρθρου 21 της οδηγίας και τα συμπεράσματα σχετίζονται με την επίτευξη των στόχων της οδηγίας. Αν και υπάρχουν πολλές προκλήσεις, οι προκλήσεις δεν αφορούν την αλλαγή του νομικού πλαισίου. Πρέπει να βελτιώσουμε πολλά σημεία της θέσης εφαρμογή, εναρμονισμένα στοιχεία, συλλογή στοιχείων, μικρότερες προθεσμίες ε, για την έγκριση των προϊόντων και καλύτερη εποπτεία. Θα πρέπει να συνεργαστούμε με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ε, βιομηχανία, ε, ενώσεις περιβάλλοντος και κράτη-μέλη. Τα προϊόντα αυτά που έχουν έμεση επίπτωση στην, ε, ε, στον τομέα της ενέργειας θα μπορούσαν να ενταχθούν σε αυτή την έκθεση. Όμως, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη προϊόντα τα οποία κατασκευάζονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να δοκιμαστούν. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο αποφασίσαμε να κρατήσουμε το εύρος και το πεδίο εφαρμογής ε, της οδηγίας δεν μπορέσαμε να ε, εγκρίνουμε ορισμένα σημεία της οδηγίας Eco Design, διότι η περίοδος που είχαμε στη διάθεσή μας ήταν πολύ περιορισμένη. Θα πρέπει λοιπόν να ε, αναθεωρηθεί η οδηγία για την σήμανση προϊόντων ενέργειας που θα γίνει μέχρι το 2014. Ως προς το ε, πρόγραμμα εργασίας 12-14, φέρει δύο μέρη. Αφενός έχουμε τον κατάλογο των καταπροτεραιότητα προϊόντων και από την άλλη πλευρά τις βελτιώσεις που θα πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή και που είναι απότοκες του προηγούμενου σχεδίου. Το πρόγραμμα εργασίας εγκρίθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου του 12, που αφορά το 12-14 και ορίζει τα καταπροτεραιότητα προϊόντα ε, και την αποστήμηση της Κομισιόν μέχρι το 2014. Επίσης, τα προσβελτίωση σημεία μετά από την κατάρτιση του σχεδίου. Θα προσδώσουμε μεγάλη σημασία στο νομοθετικό σκέλος κατά προτεραιότητα και τη συνεισφορά των υπηρεσιών της Επιτροπής στη διαδικασία τυποποίησης. Ξέρω ότι η Επιτροπή Περιβάλλοντος θα επιθυμούσε να χρησιμοποιήσουμε την ε, αυτή την οδηγία Eco ε, Conception και για τις ε, βρύσες μπάνιου. Νομίζω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τα προϊόντα που σχετίζονται με την κατανάλωση ύδατος και αυτό θα το δούμε μαζί με τις εργασίες της Ίσπρα. Θα πρέπει λοιπόν να βελτιώσουμε τον κονισμό για τέτοια προϊόντα οι προπαρασκευαστικές μελέτες για τους καυστήρες ατμού, για τα παράθυρα και τις, τα εφή προϊόντα, τα εφή μηχανήματα, θα ε, ε, εκπονηθούν τις επόμενες εβδομάδες. Θα πρέπει να μην υπάρχουν ε, αντιφάσεις, ιδιαίτερα για τα παράθυρα και τα προϊόντα μόνωσης, έτσι ώστε να προβούμε σε εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε ευφυείς ε, με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Θα ήθελα να σας πω ότι τα τρία επόμενα έτη θα είμαστε πολύ απασχολημένοι. Θα πρέπει να εγκρίνουμε 20 κανονισμούς περίπου και να, να αναθεωρήσουμε αρκετούς για να βελτιώσουμε την εποπτεία της αγοράς και τη διαδικασία τυποποίησης. Αυτό θα γίνει μόνο αν συνεργαστούμε και βασίζομαι στην υποστήριξη της Επιτροπής Περιβάλλοντος για όλες μας τις δράσεις στον τομέα αυτό. Ευχαριστούμε κύριε Πετνέλη. Δύο ακόμη εκπροσώπους κομισιών έχουμε, στους οποίους θα δώσω τον λόγο, αν θέλετε. Θέλετε? Καλώς. Ξεκινάμε τότε με τους δύο συναδέλφους. Ξεκινάμε τη συζήτηση. Ο Πέτερ Λίζε έχει τουλάχιστον 10 λεπτά χρόνο ομιλίας. Και μετά ο Πάβελ. Πέτερ. Δεν θέλω να μιλήσω 10 λεπτά. Γιατί πρέπει να τοποθετηθεί η Κομισιόν επί των λεπτομεριών πριν ε, κάνουμε άλλες ερωτήσεις. Θεωρώ πως η οδηγία οικολογικού σχεδιασμού είναι πολύ σημαντικό μέσο και θεωρώ πως έχει αποδείξει την αξία της. Έχουμε μεγάλες δυνατότητες εξοικονόμησης και στις περισσότερες περιπτώσεις δεν επηρεάζεται ο καταναλωτής. Μόνο μια τεχνική εξέλιξη του προϊόντος υπάρχει. Και είναι σωστό αυτό. Θεωρώ πως ε, υποτιμάται συχνά ε, σε αντίθεση με άλλα μέτρα κλιματικά πως ο οικολογικός σχεδιασμός αφορά όλους όσους ε, σχεδιάζουν για την ευρωπαϊκή αγορά. Δηλαδή κάποιοι συνάδελφοι λένε συνεχώς το θέμα του αποτυπώματος άνθρακα και το πώς ε, θα αξιολογούμε τις αγωγές για το εάν είναι φιλική, φιλικές προς το κλίμα ή όχι. Νομίζω πως ε, ο σχεδιασμός αυτός είναι πάρα πολύ καλός γιατί μετράει αυτά τα οποία έρχονται στην ε, ευρωπαϊκή αγορά και βεβαίως τα χαρακτηριστικά αυτά είναι πολύ εντονότερα σε ευρωπαϊκά από ό,τι σε κινέζικα, αμερικάνικα κλπ. προϊόντα. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό γιατί ανησυχούσαμε πάρα πολύ καιρό γιατί το ότι το πρώτο μέτρο το οποίο είχαμε θέσει ως προτεραιότητα στην συναπόφαση όταν το 2005 είχαμε την πρώτη οδηγία οικολογικού σχεδιασμού ότι θα περιμέναμε ε, πάρα πολύ γιατί είχαμε καθυστερήσει ήδη και ε, ακούω επιτέλους πως ε, επιτέλους έχουμε τα πρώτα μέτρα ε, είναι στον τομέα της ε, θέρμανσης και το άλλο αφορά το ζήτημα του ζεστού νερού. Και θα θέλαμε να μάθουμε ποια είναι αυτά τα μέτρα του Κομισιόν. Εδώ πέρα υπάρχει βεβαίως μια δίκαιη αντίρρηση όσον αφορά το εμπόριο από το διαδίκτυο, γιατί ε, μέχρι τώρα τα αυτοκόλλητα της ενεργειακής απόδοσης δεν μπορούσε κανείς να τα δει στο διαδίκτυο. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω από την Κομισιόν εδώ πέρα κάποιε λεπτομέρειες. Κατόπιν ο κύριος Διευθυντής είπε πως η Επιτροπή θέλει να ρυθμίσει τα τηλέφωνα του ντους και τις βρύσης. Κάποιοι συνάδελφοι το επιθυμούν, αλλά εμείς ως ΕΛΚ δεν το επιθυμούμε. Το θεωρούμε επικίνδυνο εγώ υποστηρίζω την οδηγία οικολογικού σχεδιασμού. Α, μην ξεχνάτε όμως ότι είχαμε δώσει αγώνα και για, τις, ε, για τους λαμπτήρες πυρακτώσεως, αλλά ε, τελικά χάσαμε το παιχνίδι στην επικοινωνία και στις λεπτομέρειες. Και με τα ντους και τα υπόλοιπα θα έχουμε ακόμα ένα πρόβλημα. Ντους και βρύσες, που δεν το είχαμε με τους λαμπτήρες πυρακτώσεως, δεν υπάρχει ενιαία ευρωπαϊκή σήμανση για αυτά τα δύο προϊόντα. Και πρέπει πρώτα να γίνει αυτό για μερικά χρόνια και να μπορεί εθελοντικά ο καταναλωτής να διαλέξει πιο οικονομικά τηλέφωνα τους. Δεν πρέπει να περάσουμε σε απαγορεύσεις. Οπότε... Ε, έχω συνομιλήσει και με τον Ρίχαρτ Τζέμπερ και τα λοιπά, μπορώ να σου πω, εμείς δεν θέλουμε κάτι τέτοιο. Δείτε αν υπάρχει κάποια πλειοψηφία, αλλά δεν είναι σωστό ε, να λέμε πως το θέλει η ε, Επιτροπή Περιβάλλοντος. Σας επικεντρωθούμε σε αυτά τα οποία θέλουμε και δεν επηρεάζουν τους καταναλωτές. Τον είναι κάτι διαφορετικό, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Το τηλέφωνο του ντους. Και οι κατασκευαστές μας λένε άμα κάνετε ε, και να το κάνετε αναγκαστικά θα, θα, θα, θα το κάνουν μόνοι τους οι καταναλωτές, θα το ανοίξουν και δεν θα λειτουργεί ούτως ή άλλως όπως θέλετε. Ας βάλουμε την ετικέτα και δεν χρειάζεται ρύθμιση. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε Πέτερ Λίζη. Pavel Pok. Děkuji, pane... No, pardon. Eh, děkuji, pane předsedo. Ευχαριστώ, Presidente. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συγγνώμη. Η οδηγία αυτή είναι πολύ χρήσιμη για τους καταναλωτές. Θα ήθελα να σχολιάσω το θέμα της σήμανσης ε, ηλεκτρονικών υπολογιστών και γενικότερα εξοπλισμού πληροφορικής. Ε, ποια είναι η γνώμη της Κομισιόν γι' αυτό. Το θέμα αυτό καλύπτεται από, από τον τύπο στην, στη χώρα μου, στην Τσεχική Δημοκρατία, ακούστηκαν πολλές αντιρρήσεις για το θέμα της σήμανσης των, του εξοπλισμού πληροφορικής. Ε, άλλη ερώτηση είναι εξής. Έχετε ολοκληρώσει την... Έχετε ολοκληρώσει την αξιολόγηση του εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας. Μάλιστα. Τώρα θα θέλαμε να μας πείτε και κάποια πράγματα για την κατάταξη των ηλεκτρικών σκουπών. Και ο Πέτερ Λίζε την προηγούμενη εβδομάδα μίλησε για την αποτελεσματικότητα. Γιατί οι καταναλωτές αυτό κοιτάνε και αναμένουν όταν μιλάμε για μια κατάταξη των προϊόντων. Αν λοιπόν ε, έχω μία σκούπα με λιγότερα βατ ε, ε, και ένα ωραίο ευρωπαϊκό προϊόν με πέντε βούρτσες εκεί πέρα που κάνει, καθαρίζει το χαλί μου. Αλλά τι θα δει ο καταναλωτής όταν δει τα λιγότερα βάτ, θα σκεφτεί ότι δεν είναι εξίσου αποτελεσματική η μία σκούπα με την άλλη. Οπότε, πώς θα αξιολογήσετε και θα κατατάξετε την αποτελεσματικότητα της ηλεκτρικής σκούπας. Δηλαδή, μετράτε, μετράτε το αποτέλεσμα ή κοιτάτε το μόνο την ε, κατανάλωση του ηλεκτρισμού σε σχέση με την απόδοση. Γιατί... Ε, δεν ξέρω. Κι εγώ, κι εγώ μηχανικός είμαι. Κοίταγα εκεί πέρα τους τύπους που έχετε γράψει και δεν καταλαβαίνω πώς, πώς φτάνετε σε αυτά τα αποτελέσματα που γράφετε κάτι 0,2 όσον αφορά την αφαίρεση της κόνης κτλ. Το... Λοιπόν, Κομισιόν και μετά Λίζε και μετά ΠΟΚ. Είμαι ο Πολ Χόψον από τη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας. Ε, καλωσορίζουμε και εμείς αυτή την ομοθεσία. Θα ήθελα να καθισχάσω τον κύριο Λίζε. Ο, πράγματι καθαρίζουμε όλα αυτά τα, ε, αυτές οι κρεμότητες που είχαν μείνει ο τελευταίος μήνας ήταν ε, μήνας θαυμάτων θα έλεγα, γιατί οθετήσαμε νομοθεσία και για τις ε, σκούπες και για τους ε, υπολογιστές. Στο τέλος του περασμένου μήνα συγκεκριμένα. Την περασμένη εβδομάδα, μετά από 7 χρόνια, υιοθετήσαμε και ελάχιστες απαιτήσει για boilers, εξοπλισμό θέρμανσης δηλαδή, 40-45 εκατομμύρια τόνοι ισοδύναμου πετρελαίου εξοικονομούνται έτσι. Και ε, αν όλα πάνε καλά, σήμερα το απόγευμα θα υιοθετήσουμε και άλλο ένα κείμενο για να καλύψουμε και τις ε, ε απαιτήσει stand-by και για τα δίκτυα. Ελπίζουμε ότι όλα αυτά τα κείμενα θα τα δεχτείτε και θα τα υποδεχτείτε πολύ θετικά. Εσείς και το Συμβούλιο. Και έχουμε και άλλα, για παράδειγμα τη σήμανση του δικτύου, του ίντερνετ, συγγνώμη, ηλεκτρικούς και βιομηχανικούς κινητήρες ε, και αφού τελειώσαμε με τους boilers θα περάσουμε και στους boilers με, με στερεά καύσιμα Και έχουμε και το θέμα των grills. Κουζίνες. Ηλεκτρικές κουζίνες και μάτια ηλεκτρικών κουζίνων. Ε, δεν γνωρίζω το θέμα που προέκυψε στην Τσεχική Δημοκρατία. Ομολογώ ότι δεν το γνωρίζω, να το δούμε. Αλλά η νομοθεσία που υιοθετήσαμε για τους υπολογιστές ε, είναι, αφορούν ελάχιστες απαιτήσει και χρησιμοποιούμε το πρόγραμμα Energy Star των ΗΠΑ για την σήμανση των υπολογιστών. Έχουμε ευθύνη να λειτουργεί σωστά, αλλά δεν καλύπτεται το θέμα αυτό από τις νομοθεσίες που υιοθετήσαμε πρόσφατα. Σε ό,τι αφορά το θέμα της, ε, των, της ηλεκτρικής σκούπας ε, που έθεσε ο πρόεδρος, πράγματι υπήρχε μια ανησυχία. Πρέπει να κάνουμε κάτι για τις ηλεκτρικές σκούπες, γιατί χωρίς ελάχιστες απαιτήσει οι κατασκευαστές λένε ε, ότι ε, όσο περισσότερη ενέργεια καταναλώνει μια σκούπα τόσο καλύτερα καθαρίζει. Αυτό δεν είναι, Δεν είναι σωστό. Ε, η πρότασή μας επέτρεπε ηλεκτρικές σκούπες που έχουν χαμηλή καταναλωσή και χαμηλή ισχύ απορρόφησης να παίρνουν καλή βαθμολογία. αυτό ήταν από τα αποτελέσματα της πρότασής μας αυξήσαμε τον παράγοντα αυτό από το 0,5 στο 0,2, από ε, το 0,15 στο 0,20 ε, αυτό το συντελεστή και ε, ε φέραμε πιο νωρί την πλήρη απαγόρευση των μη αποδοτικών ε, σκουπών. Ε, δεν θα μπορούν να τίθενται σε κυκλοφορία στο μέλλον τέτοιου είδου ηλεκτρικέ σκούπες. Η Επιτροπή ΙΤΡΕ ελπίζω ότι θα αναγνωρίσει πω αυτό είναι ε, το σωστό βήμα. Να δώσω το λόγο και στον κ. Μίσιγκερ για την, από τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντο. Yes, I would like to address the question... Ε, να αναφερθώ στα προϊόντα νερού. Να τονίσω πως η κατηγορία αυτή των προϊόντων συμπεριελήφθη στο πρόγραμμα εργασίας 2012-2014 με βάση μελέτες που ήταν διαθέσιμες και εξέταζαν την δυνατότητα εξοικονόμησης και ενέργειας και νερού. Οι οικονομίες αυτές είναι σημαντικές, παραδείγματο χάρη η δυνατότητα εξοικονόμησης ενέργειας είναι γύρω στα 900 γιγατζάουλ το έτος. Ε, πρέπει δηλαδή μιλάμε για τη συνολική κατανάλωση ρεύματος της Ρουμανίας το 2010 ή 54 ηλεκτρικά μέσα ηλεκτρικά εργοστάσια. Και είναι το προϊόν το οποίο μας δίνει την δεύτερη μεγαλύτερη δυνατότητα εξοικονόμησης ενέργειας από τα προϊόντα που δεν έχουν ακόμα ε, καλυφθεί από την οδηγία οικολογικού σχεδιασμού. Μιλάμε δηλαδή για μια δυνατότητα, για ένα ποσό που φτάνει μέχρι το 40% της οικιακής κατανάλωσης νερού στην Ευρώπη, από 4 έως 40% κυμαίνεται, Και θέλω να τονίσω πως ε, το γεγονός πως ε, συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα εργασίας δεν σημαίνει πως ε, έχει αποφασιστεί πως θα έχουμε κάποια εφαρμοστικά μέτρα. Αντιθέτως, τι σημαίνει. Η Εκομισιόν θα κάνει περισσότερες μελέτες που θα εξετάσουν λεπτομερώς τις πιθανές οικονομίες και θα δουν και το καλύτερο μέτρο πολιτικής για να επιτύχουμε την υψηλότερη εξοικονόμηση. Είτε λοιπόν μπορεί να είναι μια τέτοια απόφαση, μπορεί να είναι σήμανση ή εθελοντική συμφωνία της βιομηχανίας. Αυτό το οποίο σκοπεύουμε να κάνουμε λοιπόν τους επόμενους τα επόμενα ένα-δύο χρόνια είναι να δούμε την όλη κατάσταση. Θα εξετάσουμε και την ε, ικανοποίηση του πελάτη βεβαίως. Το τεχνολογικά εφικτό γνωρίζουμε πως υπάρχουν ήδη κάποιες λύσεις που δίνουν την ίδια ικανοποίηση του καταναλωτή. Υπάρχουν στην αγορά, είναι φτηνά. Η απόσβεση αυτής της τεχνολογίας διαρκεί 1 έως 20 μήνες, ενώ το προϊόν διαρκεί 15 ε, με 20 χρόνια. Οπότε είναι πολύ φτηνή η λύση. Αλλά οι μελέτες θα αξιολογήσουν όλες αυτές τις πτυχές και μόνο αφού ολοκληρωθούν οι μελέτες θα προτείνει η Κομισιόν ε, ανάλογα μέτρα, τα οποία βεβαίως θα εξετάσει το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίαση αυτή. Ο Πέτερ Λίζε έχει άλλη μια ερώτηση. Ναι. Για τις κεφαλές του Ντούς και τις Βρύσες. Να απευθύνω έκκληση. Το συντομότερο δυνατό να έχουμε σήμανση και καμία αρρύθμιση θεωρώ σε πρώτη φάση. Είναι σημαντικό να αφήσουμε λίγο χρόνο να δράσει η η σήμανση. Τα νούμερα τα οποία είπατε, ο δεύτερος μεγαλύτερος δυνατός αντίκτυπος των προϊόντων με τα οποία δεν έχουμε ασχοληθεί, ποια είναι η τάξη μεγέθους και ποιο είναι το προϊόν το οποίο θα μπορούσε να έχει τον μεγαλύτερο αντίκτυπο. Έτσι για να έχουμε και μια αίσθηση του, των μεγεθών. Μετά, το ζήτημα για τους λέβητες θερμοσύφωνες Πράγματι θα το δούμε, αλλά θεωρώ πως μετά από τόσα χρόνια Δεν ξέρω, θα μπορούσαμε να ζητήσουμε και την απόρριψη του, της πρότασης, αλλά θέλω μία εξήγηση. Γιατί πρότεινε κάτι τέτοιο η Κομισιόν, ποια διαφορετικά επιχειρήματα έπαιξαν ρόλο. Το ίδιο και για το νερό, το ζεστό νερό. Και το ίδιο θα ήθελα να μάθω για τα προτινόμενα μέτρα. Άκουσα κάτι για ηλεκτρικούς κινητήρες. Νομίζω το είχαμε καλύψει. Ήταν το μεγαλύτερο μέτρο που υπήρχε μέχρι στιγμής. Αλλά θα ήθελα να καταλάβω καλύτερα τι έχει ρυθμιστεί, τι πρέπει να ρυθμιστεί ακόμα και για το θέμα κουζίνες, γκριλ και τα λοιπά. Και αυτό το θέμα πρέπει να το δούμε. Για να μην ε, υπάρξει πάλι καμία θύελα της κοινή γνώμης και δεν μπορούμε να αντιδράσουμε. Μάλιστα. Θα ήθελα και εγώ να συμπληρώσω το εξής. Έχουμε μεγάλο φίλος του οικολογικού σχεδιασμού. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο δυναμικό εξοικονόμησης και μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα για να πάμε σε μια πιο αποτελεσματική έτσι, κοινότητα. Αλλά το θέμα είναι όταν ακούμε κάποιες λέξεις, δηλαδή όταν ακούμε τη λέξη grill. Έχω περάσει κάποια χρόνια εδώ μέσα Κοιτάξτε, υπάρχουν εδώ πέρα όταν θα πάμε προς τις ευρωεκλογές πάρα πολύ πονηροί συνάδελφοι και σας παρακαλώ να το σκέφτεστε και αυτό στην Κομισιόν πως ορισμένα πράγματα προσφέρονται για σλόγγαν, έτσι, για συνθήματα. Να σκέφτεστε λοιπόν πώς θα διαμορφωθεί η επικοινωνία ορισμένων πραγμάτων. Έτσι. Για τον ντους, παραδείγματο χάρη, για τις βρύσεις. Ακούγονται διάφορες τερατολογίες. Βγείτε και ξεκαθαρίστε το. Δεν ε, σκοπεύουμε να κάνουμε τίποτα. Ή Στη δική μου την ε, περιοχή, παραδείγματο χάρη, υπάρχει το πρόβλημα ότι χρησιμοποιούν πάρα πολύ λίγο νερό και δεν λειτουργούν σωστά οι σωλήνε. Και η εταιρεία ίδρυυση αναγκάζεται ε, να ανεβάζει την πίεση και να του λέει ε, τραβήξτε λίγο περισσότερο νερό για να ξεμπλοκάρουν οι σωλήνε. Πρέπει δηλαδή και να το δούμε και αυτό το πράγμα. Και εσεί να προσέξετε ιδιαίτερα του επόμενου μήνε, σα παρακαλώ το θέμα τη επικοινωνία. Λοιπόν, τον λόγο έχει πάλι η Κομισιόν. Ποιο θέλει να μιλήσει. Uh, uh, Ίσως να σας δώσω κάποια στοιχεία καταρχήν για τον πραγματικό αντίκτυπο των μέτρων μας και μετά θα δώσω το λόγο στους υπόλοιπους συναδέλφους να απαντήσουν σε πιο συγκεκριμένα ζητήματα. Ε, ο, το εκτιμόμενος αντίκτυπος για τα προϊόντα ύδατος, όπως βρύσες κλπ, ε, που είναι το νούμερο ένα στη λίστα μας, είναι 885 γιγατζάουλ το χρόνο. Δεύτερο στη λίστα, ε, οι ευφυείς μετρητές, 802 ε, πέτατζάουλ και τρίτον, προϊόντα της οικοδομής, 785 πέτατζάουλ το χρόνο για τα παράθυρα τα προϊόντα μη που δεν προτεραιότητας, ε, η θερμομόνωση, από αυτά η θερμομόνωση είναι το πιο σημαντικό, 1500 πεντατζάουλ το χρόνο. Το άδω στο λόγο συναδέλφους. Ο κ. Λίζε ρώτησε για τους φούρνους, τα μάτια, και τα γκριλ και για τους ηλεκτρικούς κινητήρες. Είναι μια μικρή τροπολογία, αλλά δυστυχώς δεν γνωρίζω ποια είναι. Ε, θα σας ενημερώσω. Ε, ε, καταλαβαίνω βέβαια εν γέννη ότι ορισμένα από αυτά είναι θέματα πολύ σημαντικά. Πολύ ευχαρίστω να σας δώσουμε πληροφορίες ε, είτε στην Επιτροπή είτε Σε ό,τι αφορά τις πωλήσει ε, είναι κρίσιμο. Ε, η θυσιότητα αφορά την επικοινωνία είναι πολύ κρίσιμο θέμα. Ε, έχετε δίκιο, λέω. Ε, ένα όμως από τα πιο, μία από τι πιο ε, αναγνωρισμένες ε, πολιτικές Ευρωπαϊκή Ένωση Ένωσης είναι αυτή. Ε, αν πάτε σε ένα πάρτι και ρωτήσετε, σας ρωτήσουν τι κάνετε και τους πείτε εγώ βάζω τις ετικέτες ενεργειακής απόδοσης στα ε, πλυντήρια ε, ή στα ψυγεία, α, β, σε κατηγορία κλπ. Ε, πολύ πρόσφατα έχουν αρχίσει και αναγνωρίζουν τι κάνω. Είναι νομίζω ένας τομέας πολιτικής που πραγματικά έχει φτάσει στους πολίτες μας και έχει αναγνωριστεί η προσπάθειά μας. Να απαντήσω στο ερώτημα τη σήμανση και προτεραιότητα για τη σήμανση, για τα προϊόντα ύδατο. δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να προδικάσουμε ποιες είναι, ποια είναι τα καλύτερα μέτρα για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατηγορία προϊόντων. Ούτε και ποια είναι για να πάρουμε τα καλύτερα, τα περισσότερα ωφέλη. Έχουμε εμπειρία με την εφαρμογή τη οδηγία Eco Design. Ε, μόνο στο τέλος των ε, μελετών προετοιμασίας μπορούσαμε να πούμε ε, ποια είναι πιο σωστή επιλογή και πάντοτε, μα συνήθως, ε, τα ελάχιστα, οι ελάχιστε απαιτήσει μαζί με την σήμανση, ένα καλό μείγμα αυτών των δύο είναι συνήθως, τις περισσότερες φορές, η καλύτερη λύση. άλλες φορές βέβαια υπάρχει και εναλλακτική λύση της ε, συμφωνίας ε, ε, μεταξύ των κατασκευαστών, της δέσμευσής τους δηλαδή. Γι' αυτό το δούμε αφού γίνουν μελέτες. Τώρα, σε ό,τι αφορά το αποτέλεσμα της μείωσης της χρήσης νερού στα νοικοκυριά την, ε, το σχεδιασμό των συστημάτων των δικτύων αποχέτευσης και τα αποτελέσματά του κλπ. Κάναμε κάποιες πρώτες μελέτες και δεν βρήκαμε αποδείξεις ότι η, μειω... <coughs> η μειωμένη χρήση νερού θα έχει αρνητικές συνέπειες στα, στα δίκτυα αποχέτευσης. Αλλά ακόμα και αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, είμαστε ε, πεπισμένοι ότι ε, ο καθαρισμός των δικτύων αποχέτευση δεν πρέπει να γίνεται με ζεστό νερό ή με πόσιμο νερό, αλλά με ε, νερό που έχει χαμηλότερες, λιγότερες βλαπτικές συνέπειες για το περιβάλλον. Επίσης, δεν θα πρέπει να πληρώνουν οι, καταναλωτές μέσω των ε, συνήθων χρεώσεων κατανάλωση νερού για τον καθαρισμό των αποχετεύσεων του δικτύου αποχετεύσεως. Θα πρέπει να μελετήσουμε ακόμα περισσότερο βέβαια τα θέματα αυτά στις ε, ε, μελέτες μας και όταν έχουμε περισσότερα στοιχεία στα χέρια μας θα μπορέσουμε να προτείνουμε την καλύτερη λύση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. μα Πέτερ Λίζε, έβδομη φορά παίρνει το λόγο. Ε, ναι, είναι που έχουμε χρόνο σήμερα. Λοιπόν, Μία ερώτηση έχω στον κύριο που ανέφερε τα 7 μέτρα για τα 7 χρόνια, με συγχωρείτε, το διάσημο αυτό μέτρο για τους καυστήρες και τους ε, Τώρα, Είχαμε αυτή τη συζήτηση για τη σήμανση αν θα είναι πράσινο, κίτρινο, κόκκινο ή αν θα είναι α, α συν και τα λοιπά. Και το ερώτημα ήταν αν θα το βάζει ο κατασκευαστής ή ο εγκαταστάτης ο οποίος το προσαρμόζει αν θα έχει τη δυνατότητα να βάλει ένα αυτοκόλλητο επιτόπου. Και είπατε πως κάποιοι μη αποτελεσματικοί οι τέτοιοι λέβητες δεν θα επιτρέπονται πλέον. Θα ήθελα να μάθω λοιπόν μετά από όλα αυτά, μετά από όλη αυτή η δικασία των 7 ποιος ήταν ο συμβιβασμός που επέτρεψε να προχωρήσουμε. Ναι, εδώ, εδώ είμαι. Και να δώσω το λόγο. Άλλο συνάλφος δεν έχει ε, άλλη ερώτηση. Για τις βρύσες είπατε 158 πετατζάουλ για τις βρύσες. 158 ή λάθος έγραψα. Η Κομισιόν. Ποιος θέλει να απαντήσει. 885. Εντυπωσιακό. Μάλιστα. Κύριε Χέρτσεν. Να με συγχωρείτε κύριε Πρόεδρε για να απαντήσω στον κύριο Λίζε. Ο κανονισμός για τις ετικέτες για την θέρμανση το 2015 θα είναι α, α συν και α2 συν. Η συζήτηση είναι πάμε σε α και 3 συν και η συμβαστική πρόταση είναι να πάμε σε α τρία συν, αλλά μόνο μετά από μια αναθεώρηση. Και το ερώτημα είναι, το α, όπως ξέρουμε, είναι η καλύτερη επίδοση που μπορεί να επιτευχθεί από καυστήρες ορεκτών καυσίμων από μόνος τους. Δηλαδή για να το ξεπεράσουμε πρέπει να υπάρξει είτε μία ε, μικρό συμπαραγωγή, είτε αντλία θερμότητας, είτε κάτι ηλιακό. Θα παραμένουν λοιπόν ως πράσινοι στο χρώμα μέχρι η αναθεώρηση να δείξει το εάν έχουμε αρκετά φτηνές εναλλακτικές που θα επιτρέψουν να πάμε πιο πάνω το φάσμα. Αυτό ήταν ο συμβιβασμό. Τώρα για τον εγκαταστάτη, για το ποιο θα βάλει την ετικέτα. Το αποτέλεσμα ήταν είτε ο εγκαταστάτη είτε ο κατασκευαστή. Μπορεί να βάλει την ετικέτα στο σύστημα. Δηλαδή, ένα κατασκευαστή που έρχεται με ένα ολόκληρο σύστημα μπορεί να το πουλήσει με την ετικέτα. Αλλιώ, ο εγκαταστάτη που θα φτιάξει ένα σύστημα με διαφορετικά στοιχεία θα βάλει την ετικέτα. Για τον οικολογικό σχεδιασμό δεν είχαμε σημαντικές αλλαγές σε σύγκριση με την πρόταση που υπάρχει εδώ και ένα έτος, οπότε θα έχουμε κάποιες προδιαγραφές μετά από ένα έτος, ένα, κάποιες δεύτερες μετά από τέσσερα χρόνια και μετά από πέντε, μετά από αυτό. Η κύρια αλλαγή η οποία έγινε σε ελάχιστες προδιαγραφές για ε, καυστήρες και θερμοσύφωνες ε, αφορούσε εκπομπές ε, μονοξιδίου του αζότου οι οποίες θα επιβληθούν αργότερα αλλά θα είναι αυστηρότερες γιατί κάποιες χώρες έχουν ήδη κάποιες ε, προδιαγραφές. Οπότε επειδή δίνουμε πέντε χρόνια αντί για τρία στους κατασκευαστές, δίνουμε στους κατασκευαστές το ε, περιθώριο να επιτύχουν αυτό το αποτέλεσμα. Και στις χώρες που δεν έχουν αυστηρές προδιαγραφές. Αυτές είναι οι αλλαγές στην πρόταση που θα σας ε, στείλουμε. Ευχαριστώ. Νομίζω πως έχουν απαντηθεί όλες οι ερωτήσεις. Εξακολουθήσατε, λοιπόν, στον δρόμο για μια πιο αποτελεσματική χρήση ενέργειας. Τα νούμερα μιλάνε από μόνα τους. Να δούμε τα νούμερα δηλαδή αντιστοιχούν πραγματικά σε ολόκληρα ηλεκτρικά εργοστάσια και είναι εντυπωσιακό. Δηλαδή η ενέργεια που δεν καταναλώνει κανείς νομίζω είναι το καλύτερο που μπορεί να κάνει ο νομοθέτης. Και σας παρακαλώ ακόμη μια φορά προσέξτε το θέμα της επικοινωνίας γιατί πλησιάζουν και ευρωεκλογές και γινόμαστε και πιο νευρικοί καταλαβαίνετε. Ευχαριστώ λοιπόν ιδιαίτερα την Κομισιόν για την ε, καλή αυτή παρουσίαση. Ήταν πάρα πολύ χρήσιμη. Σας ευχαριστώ. Περνάμε στο επόμενο θέμα της ημερησίας διάταξης. Το θέμα εδώ είναι ο θόρυβος. Το τμήμα πολιτικής θα μας κάνει είχαμε παρουσιάσει μια μελέτη που είχαμε ζητήσει να γίνει, γιατί το θέμα του θορύβου δεν έχει ερευνηθεί αρκετά και δεν παίζει τόσο μεγάλο ρόλο στην πολιτική του περιβάλλοντος, αλλά στην πολιτική υγείας. Έχουμε λοιπόν μια νομοθετική διαδικασία και το θέμα αφορούσε την στάθμη θορύβου των ε, οχημάτων, αλλά ο θόρυβος και ο ήχος ε, παράγεται και από άλλες πηγές. Τρένα, αεροπλάνα και νομίζω πως ε, μπορούμε να ασχοληθούμε και με αυτό το θέμα της δημόσιας υγείας και από μια έτσι επιστημονικά θεμελιωμένη ε, σκοπιά να το αξιολογήσουμε. Παρακαλώ λοιπόν να μας κάνετε την παρουσίαση. Ποιος ε, θα ξεκινήσει, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Καλό σας απόγευμα. Θα σας παρουσιάσω τα βασικά μηνύματα, τα αποτελέσματα μιας μελέτης της Μιλιέ προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που φέρει τον τίτλο «Προς μία ολοκληρωμένη στρατηγική για το θόρυβο». Η συγγραφής είναι η Μόνικα Γκουαρινόνη και εγώ η Κάθριν Γκάνσλεϊμ. με τη βοήθεια του, ενός ακαδημαϊκού του κυρίου Μέρφη. Θα σας μιλήσω για τις πηγές έκθεσης στον περιβαλλοντικό θόρυβο. Θα σας μιλήσω για τις επιπτώσεις στην υγεία, το νομοθετικό πλαίσιο, την ε, βασική νομοθεσία και τις πρόσφατες εξελίξεις, καθώς και την προστιθέμενη αξία της περαιτέρω δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση του θορύβου. Αρχίζοντας ε, με, από τις πηγές έκθεσης, οι βασικές πηγές αφορούν τις μεταφορές ε, τις κατασκευαστικές εταιρείες, τη βιομηχανία, τα μπαρ, τους γείτονες, πηγές αναψυχής, από κέντρα αναψυχής και από το σπίτι. Τώρα θα αναφερθώ στις μεταφορές, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα. Τα στοιχεία αυτά που βλέπετε στη γραφική αυτή παράσταση είναι τα στοιχεία τα οποία υποβλήθηκαν δυνάμει της end το, του 2007, δηλαδή της οδηγίας αντιμετώπισης του περιβαλλοντικού ε, θορύβου. Με μπλε σκιαγραφούνται εκείνοι οι οποίοι εκτίθενται στο θόρυβο κατά τη διάρκεια της ημέρας και το βράδυ, πάνω από 55 δεσιμπέλ, ενώ σε κόκκινο βλέπετε ποιοι εκτίθενται στο θόρυβο από τις μεταφορές τη νύχτα πάνω από 50 δεσιμπέλ. Και εδώ έχετε τους δείκτες που υπάρχουν στην οδηγία. Βλέπουμε λοιπόν ότι μία πρωτογενής πηγή θορύβου και την ημέρα και τη νύχτα είναι οι οδικές μεταφορές. Μιλάμε για 26 εκατομμύρια 56 εκατομμύρια που εκτίθενται σε θόρυβο πάντα από 55 δεσιμπέλ ημερησίως. Υπάρχει και μία έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος του 8 που δείχνει ότι το 55% εκείνων που κατοικούν σε αστικές περιοχές εκτίθενται σε θόρυβο περίπου 55 δεσιμπέλ έχετε πολύ χαμηλότερα στοιχεία σε σχέση με τις σιδηροδρομικές μεταφορές, αεροδρόμια και ε, βιομηχανία. Θεωρούμε πολλές φορές ότι τα αεροπλάνα είναι πιο ενοχλητικά. Βλέπουμε όμως ότι ο θόρυβος είναι πολύ ενοχλητικός παρόλο που οι δείκτες είναι σχετικά ε, χαμηλοί. Εδώ έχετε συγκρίσιμα στοιχεία εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων. Βλέπετε λοιπόν ότι η βασική πηγή θορύβου αφορά τους μεγάλους οδικούς άξονες. Τώρα, περνώντας ε, στις επιπτώσεις στην υγεία, ε, καταρχήν είναι το γεγονός της όχλησης και έχουμε στοιχεία από τον ΠΟΗ για το 2011 σε σχέση με τις ασθένειες που προκαλούνται από το θόρυβο. Βλέπουμε λοιπόν ότι μας έδωσαν μία μεθοδολογία αναφοράς και ε, είδαμε ποιες ασθένειες δημιουργούνται. Μιλάμε λοιπόν το, το πώς, υγεία, πώς υγεία μπορούμε να απολέσουμε από την έκθεση στο θόρυβο. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει η όχληση. Um, in the green. Οι διαταραχές ύπνου είναι ε, το πρώτο. Μετά είναι η όχληση. Ε, επίσης, σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία Και εδώ μιλάμε και για ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες, δηλαδή παιδιά τα οποία έχουν γνωστικά προβλήματα ή γνωστικές, γνωστικής υφής ασθένειες ή ευάλωτα άτομα τα οποία πάσχουν από καρδιακές νόσους. Το ίδιο έγγραφο του ΠΟΗ του 11 τονίζει ότι στη Δυτική Ευρώπη ένας στους τρεις πλήττεται από το θόρυβο, ένας στους πέντε έχει προβλήματα ύπνου και αυτό οδηγεί σε 1 με 1,6 ε, της 100 ε, απώλειες σε σχέση με ε, θόρυβο από τον οποίο εκτίθεται κανείς. Σε σχέση τώρα με ε, ότι με το, τη μελέτη του Ευρωβαρομέτρου ορίζει ότι το 44% θεωρεί ότι ο θόρυβος πλήττει την ανθρώπινη υγεία σε ευρύ βαθμό. Και ο ΠΟΗ θεωρεί την ηχορύπανση πολύ μεγάλη όχληση, πηγή όχλησης μετά από την ατμοσφαιρική ρύπανση. Άρα το ρυθμιστικό πλαίσιο περιλαμβάνει την οδηγία του 2 49 για την αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού θορύβου και αυτό αφορά τις ε, ε, σιδηροδρομικές μεταφορές, τις οδικές μεταφορές, τις εναέριες, ε, οχήματα, μηχανήματα κλπ. Άρα θα πρέπει να υπάρχει συμπληρωματικός χαρακτήρας έτσι ώστε να μειώσουμε την έκθεση του λήπτη με βάση την οδηγία αντιμετώπισης ε, του θορύβου από το περιβάλλον. Το 2011 λοιπόν συντάχθηκε μία έκθεση για την εφαρμογή της οδηγίας END και με βάση τα στοιχεία και την έκβαση φτάσαμε σε μια συλλογή στοιχείων και εποπτείας με βάση στρατηγικούς χάρτες και προγράμματα δράσης. Ο πρώτος γύρος έχει ολοκληρωθεί. Η δεύτερη χαρτογράφηση έπρεπε να υποβληθεί το Δεκέμβριο του 2012. Όμως το 30% της ε, χαρτογράφησης μόνο έχει ολοκληρωθεί. Η οδηγία END μας οδήγησε σε μεγαλύτερη συνειδητοποίηση του ζητήματος από πλευράς κοινού αλλά και υπαλλήλων που εργάζονται επί του θέματος και γι' αυτό δίνουμε στο θόρυβο μεγαλύτερη προτεραιότητα έτσι ώστε να υπάρξει και κατάλληλη πολιτική θέληση αντιμετώπισης. Και μιλάμε και για βέλτιστη πρακτική μεταξύ κρατών μελών. Ως προς την αποτελεσματικότητα όμως της οδηγίας αυτής της END, δυστυχώς δεν έχουμε μειώσει ε, τις επιπτώσεις του θορύβου. Είχαμε και καθυστερήσεις στην εφαρμογή, η ποιότητα της χαρτογράφησης και των προγραμμάτων δράσης δεν είναι και τόσο καλή και υπάρχουν ασυμβατότητες στη μεθοδολογία χαρτογράφησης, διότι τα κράτη-μέλη χρησιμοποίησαν διαφορετική μεθοδολογία. Άρα είναι δύσκολο να συγκρίνουμε τα αποτελέσματα της χαρτογράφησης ανά τα κράτη-μέλη και υπάρχει και σύγχυση ως προσορισμένα προαπαιτούμενα. Ως προς την πρόοδο που έχει επιτελεστεί, εγκρίθηκε μία κοινή μεθοδολογία για την αποτίμηση του θορύβου που θα οδηγήσει στην αναθεώρηση του παραρτήματος 2 της οδηγίας END και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος ζητά καλύτερη εκτίμηση και ε, καλύτερο reporting πού μπορεί να υπάρξει μεγαλύτερη πρόοδος. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να έχουμε καλύτερες κατευθυντήριες γραμμές και δυστυχώς δεν είναι υποχρεωτικό να εφαρμόζονται τα προγράμματα δράσης. Γιατί το ζήτημα είναι ελήψη κοινών στόχων ή οριακών τιμών. Για τι δέσμευση μιλάμε, τι θα επιβληθεί υποχρεωτικά. Μιλάμε λοιπόν για οριακές τιμές μέσα στα πλαίσια της οδηγίας αυτής και θέλουμε να γνωρίζουμε κατά πόσο μπορούμε να έχουμε οριακές τιμές, τιμές εκκίνησης ή τιμές στόχου. Οι εμπειρογνώμονες μας λένε ότι ο μακροχρόνιος στόχος είναι να έχουμε οριακές τιμές που να εμπεριέχονται στην ομοθεσία. Υπάρχουν και επιχειρήματα σε σχέση με την επικουρικότητα, σε σχέση με τα κράτη-μέλη που θα πρέπει να μπορούν να αποφασίζουν καθεαυτά με βάση το πολιτισμικό υπόβαθρο περί αποδοχής θορύβου. Και εάν αυτό το συνδυάσουμε με την γενική ανησυχία του κοινού, βλέπουμε ότι θα πρέπει να αναθεωρήσουμε τις οριακές τιμές. Υπάρχει και το θέμα της χαρτογράφησης θορύβου που δεν είναι συγκρίσιμη και αυτό αποτελεί μεγάλη πρόκληση γιατί αν έχουμε οριακές τιμές πώς θα τις ε, επιβάλλουμε όταν έχουμε διαφορετικές χαρτογραφήσεις. Επειδή υπάρχει διαφορά μεταξύ ε, μεθόδων υπολογισμού και μπορούμε να δούμε ποια μέθοδος χρησιμοποιείται στα κράτη-μέλη, θα πρέπει να αρκεστούμε ή να προσαρμοστούμε σε αυτό. Η επόμενη σειρά ε, χαρτογραφήσεων θα είναι συγκρίσιμη. Το 2017 και μετά δηλαδή. Σε σχέση με τις τιμές εκκίνησης, πρόκειται για τιμές κατόφλια και το οποίο θα σήμαινε ότι μετά από αυτές τις οριακές τιμές, τις τιμές εκκίνησης θα έπρεπε κανείς να δράσει ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα. Ισχύουν σε ορισμένα κράτη-μέλη και θα πρέπει ε, να λάβουμε υπόψη ότι από πολιτικής πλευράς δέχον, γίνει πιο καλά αποδεκτές αυτές οι τιμές παρά οι οριακές. Οι τιμές εκκίνησης λοιπόν είναι ευρύτερα αποδεκτές. Θα πρέπει όμως να δούμε πώς μπορούμε να ορίσουμε τον ε, ε, δεσμευτικό τους χαρακτήρα και να βρούμε και τα κατάλληλα μέσα γι' αυτό. Ως προς τις αξίες ε, στοχοθέτησης θα πρέπει να γίνουν πολιτικά αποδεκτές αλλά όταν μιλάμε για οποιασδήποτε τιμές, οριακές ή μη, θα πρέπει να τις διασυνδέσουμε με μία ε, εύρωστη νομοθετική βάση. Διαφορετικά το κόστος επίτευξης ε, έγκυται στις τοπικές αρχές και στους φορολογούμενους. Εάν δεν έχετε βασική νομοθεσία, στεναρή βασική νομοθεσία, τότε θα πρέπει να υπάρξει ελάφρυνση ε, του θορύβου σε επίπεδο αποδέκτη. Δηλαδή να ε, γίνουν αλλαγές στο συγκοινωνιακό, στα μεγάλα αστικά κέντρα. Τότε δεν πληρώνει ο ρηπαίνων, αλλά ο φορολογούμενος. Επίσης, τα μέτρα αυτά μετρίασης θα πρέπει να είναι ε, πολύ θετικά από πλευράς αποτίμησης κόστους ωφελίας ως προς τη μείωση έκθεσης ε, υψηλά δεσιμπέλ. Εάν λοιπόν ορίσουμε τιμές εκκίνησης ή οριακές ε, τιμές ή τιμές στόχου, θα πρέπει οι τοπικές αρχές να μην πρέπει να ανταποκριθούν στο κόστος. Διαφορετικά η κατάσταση θα είναι άκρος αρνητική. Άρα θεωρούμε ότι προς το παρόν δεν είναι ρεαλιστικό να ορίσουμε οριακές τιμές. Τώρα, κινούμενοι προς, προς τη βασική νομοθεσία, την πρωτογενή νομοθεσία, με βάση την έκθεση του 2012 θεωρήσαμε ότι θα πρέπει να βελτιώσουμε την νομοθεσία ως προς την εκπομπή οδικού θορύβου. Αυτή είναι πιο αποτελεσματική προσέγγιση για τον μετριασμό του θορύβου από τις οδικές αρτηρίες και θα πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι. Ως προς την πρόταση της Κομισιόν, την 2011-876 για, τα, για τις εκπομπές θορύβου από οχήματα, σε αυτό το σε αυτή την τριφασική προσέγγιση θεωρούμε ότι δεν είμαστε ιδιαίτερα φιλόδοξοι και από τεχνικής ε, πλευράς δεν έχει νόημα να τύχει υποστήριξη από την οδηγία END. Επίσης, αν λάβουμε τις αλλαγές που έχουν επέλθει από τις ε, μεθόδους δοκιμών, το πέρασμα από τη μία ε, μέθοδο στην άλλη και τη στιγμή που μιλάμε για προσωμιώσεις όταν ε, γίνονται μετρήσεις θορύβου που προέρχεται από οδικές αρτηρίες με βάση τη μέτρηση των εκπομπών οχημάτων και ιδιαίτερα όταν πρόκειται για μία διαφορά 2 δεσιμπέλ, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι μετά την έκβαση της πρώτης ανάγνωσης θα πρέπει να προσθέσουμε οπωσδήποτε δύο δεσιμπέλ σε αυτά τα στοιχεία εξαιτίας της αλλαγής στο, στη μέθοδο δοκιμών. Ως προς τη μέθοδο δοκιμών, θα πρέπει να πούμε ότι δεν λαμβάνουμε υπόψη τα ελαστικά που χρησιμοποιούνται, γιατί πολλές φορές ε, υπάρχουν ελαστικά τα οποία δεν ε, εκπέμπουν πολύ θόρυβο, και τα οποία όμως έχουν μικρό αντίκτυπο στην αγορά. Όπως την Ως προς την πρόταση της ε, Κομισιόν, είχαμε και μία μελέτη που δημοσιεύτηκε το 2012 από ένα γερμανικό φορέα, που σχετίζεται με τη μείωση εκπομπών θορύβου μέσα σε μία εικοσαετία. Μιλάμε για 1,7 δεσιμπέλ για την 20 ετία. Αυτό θα πρέπει να το λάβετε υπόψη. Ε, θα πρέπει να λάβετε υπόψη ότι για ε, τον άνθρωπο για να αντιληφθεί, αντιληφθεί τη μείωση του θορύβου θα πρέπει να είναι ανώτερη των 2 δεσιμπέλ. Μετά έχουμε την πρώτη ανάγνωση, η οποία αποδυνάμωσε περαιτέρω την πρόταση γιατί για τα βαριά οχήματα περιορίστηκε στα 81 δεσιμπέλ. Ε, αν δείτε και τις αλλαγές στις δοκιμές μπορείτε να προσθέσετε 2 δεσιμπέλ, άρα έχουν αυξηθεί ε, οι οριακές τιμές ως προς τα αυτοκίνητα σπορ γιατί για τα σπόρα αυτοκίνητα βλέπουμε ότι έχουν μεγάλη επίπτωση στις εκπομπές περιβαλλοντικού θορύβου. Υπάρχουν και άλλα μέτρα, το σύστημα οδικής ταξινόμησης που συσχετίζεται με τη χαρτογράφηση για να αναγνωρίσουμε ε, το μίσο που πρέπει να δράσουμε αλλά πάντα το κόστος μετακυλίεται στον φορολογούμενο. Επίσης, η σήμανση, η διαδικασία σήμανση ε, μετακυλεί το κόστος στον αγοραστή του οχήματος. Και επίσης έχουμε μια χρονική καθυστέρηση 6 ετών. Άρα συνολικά μπορούμε να πούμε ότι τα σχήματα αυτά δεν είναι καθόλου φιλόδοξα, οι στόχοι αυτοί και δεν οδηγούν στην σωστή εφαρμογή της οδηγίας περί περιβαλλοντικού θορύβου, της οδηγίας END. Τώρα, προχωράμε στα συμπεράσματα. Ποια είναι η προστέμενη αξία δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα θορύβου από εδώ και πέρα. Από τεχνικής πλευράς ο μετριασμός ε, του θορύβου στην πηγή είναι η πιο αποτελεσματική πλευράς κόστους στρατηγική. Όμως ε, πρακτικά υπάρχει ανάγκη ενός μείγματος πολιτικής, ε, μείωση στην πηγή και μείωση στο λήπτη. Για να βελτιώσουμε τις συνεργές ανάμεσα στη μασική νομοθεσία και την νομοθεσία END χρειάζεται μια νομοθεσία που θα, αυστηρή νομοθεσία για την θόρυβο στην πηγή. Η οδηγία ε, end όμως, ε, μάλλον ως τώρα, τα μέτρα της βασικής νομοθεσίας ε, περιθωριοποιούν σε μεγάλο βαθμό την νομοθεσία, την οδηγία end. Ε, και τελικά είναι το κόστος του φορολογούμενο θα πρέπει να συγκρίνουμε αυτή την τάση με, την, ε, με τα αποτέλεσμα του Ευρωβαρομέτρου που αναφέρουν ότι το 44% της κοινή νόμης θεωρεί πως ε, ο θόρυβος είναι ένα βασικό ε, θέμα δημόσιας υγείας. Επίσης έχουμε όλο και περισσότερες ενδείξεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τα, τις βραβερές επιπτώσεις του θορύβου στην υγεία του ανθρώπου. Ευχαριστώ. ευχαριστώ πάρα πολύ σας και τους συναδέλφους για τη σύνταξη αυτής της μελέτης. Είναι κρίμα το ότι δεν είναι εδώ πέρα συνάδελφοι σήμερα. Έχουν όλοι σοβαρούς λόγους, αλλά ήταν μια πάρα πολύ καλή εικόνα αυτή η οποία μας δώσατε για το θέμα αυτό. Ε, θόρυβος, ναι. Το θέμα δεν είναι ο λίγος θόρυβος, αλλά έχει ε, σοβαρές επιπτώσεις και για τα άτομα και για διάφορους ε, και τη, την, ε, τις κοινότητες τις διάφορες και είπατε ξεκάθαρα πως πρέπει να καταπολεμηθεί ο, πόλεμ, ο θόρυβος με συγχωρείτε στην πηγή για να μην πληρώνουν όλοι οι υπόλοιποι έτσι, με τα διάφορα μέτρα περιορισμού που δεν είναι στην πηγή. Σας ευχαριστώ. Θα μας δώσετε, ελπίζω αυτή η μελέτη και σε άλλες γλώσσες, πέρα από τα αγγλικά. Γιατί είναι καλό, γιατί δεν υπάρχουν τόσο πολλές μελέτες και γιατί η κοινή γνώμη, το παρατήρησα για τη μελέτη για το σχιστολιθικό αέριο, ε, θέλει μεταφρασμένες ε, μελέτες. Εργάστηκαν με τη δική μας μεταφρασμένη μελέτη για το σχιστολιθικό αέριο. Οπότε θα δούμε σε ποιε γλώσσε μπορούμε να τη μεταφράσουμε, γιατί νομίζω η κοινή γνώμη θα το εκτιμήσει. Η κυρία Χιούμπνερ ζήτησε το λόγο. Ναι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Με εκπλήσει ομολογώ που είμαστε τόσοι λίγοι στην αίθουσα. Ξέρουμε παρόλα αυτά ότι ένα μεγάλο ποσοστό του θορύβου δημιουργείται εκεί που ζούμε. Μας αφορά λοιπόν καθημερινά ο θόρυβο. Ε, μείωση θορύβου στην πηγή. Ε, πολύ σημαντική. Γιατί και εδώ αυτό έχει να κάνει με την καινοτομία. Είναι ένα θέμα το οποίο τονίζουμε συνεχώς. Πρέπει να είμαστε καινοτόμοι για να καταφέρουμε να μειώσουμε το θόρυβο στην πηγή. Να σας ε, επιστήσω την προσοχή σε ορισμένες λύσεις που θα μπορούσαν να υιοθετηθούν γενικά μιλήσατε για νέα ασφαλτόστρωση των δρόμων. Όταν ε, κατασκευάζονται καινούργιες αρτηρίες ή όταν κατασκευάζονται καινούργιες δρομικές γραμμές θα πρέπει να χρησιμοποιούνται οι καλύτερες ε, γνωστές τεχνολογίες και τα βέλτιστα υλικά. Προφανώ η τεχνολογία έχει βελτιωθεί σε σχέση με αυτό που ήταν πριν από 20 χρόνια. Θα πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μα. Οι ε, δρόμοι θα πρέπει να α... ανακαινίζονται, να βελτιώνονται με τη χρήση νέων υλικών. Αλλά υπάρχουν και πιο απλοί τρόποι Εγώ κοιτάω την κίνηση στις μεγάλη πόλη και βλέπω ότι θα μπορούσαμε να ε, πετύχουμε μεγάλες εξοικονομήσεις με το πράσινο κύμα στους σηματοδότες. Έτσι ώστε τα αυτοκίνητα να μην χρειάζεται να σταματάνε κάθε 100 μέτρα να περιμένουν να ανάψει πράσινο το φανάρι. Αυτό θα ε, έκανε και τα... θα αυξάνε το, τη διάρκεια ζωής ε, και των αυτοκινήτων, των οχημάτων γενικότερα και των λεωφορείων και θα μείωνε την κατανάλωση καυσίμου ε, και τις ε, εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Συνεπώς έχουμε πολλαπλά ωφέλη. Επίσης θα μπορούσαμε να Ε, δούμε ε, το θέμα της ε, επανεισαγωγής των τρόλεϊ στις πόλεις μας. Παλιότερα είχαμε πιο πολλά τρόλεϊ, ηλεκτροκίνητα μέσα μαζικής μεταφοράς στους δρόμους μας και δείχνει σαν να είναι ένα βήμα προς τα πίσω αυτό προτείνω, αλλά ίσως είναι μια καλή λύση για τις κεντρικές αρτηρίες τουλάχιστον, εκεί που παράγει το περισσότερο θόρυβος, για το κέντρο της πόλης ενδεχομένω. Στην Ελβετία, για παράδειγμα, γνωρίζω πως πολλές πόλεις ξαναφέρουν πίσω τα τρόλεϊ. Ίσως θα έπρεπε να το σκεφτούμε για τις πόλεις μας. Ε, βέβαια είναι και θέματα επικορικότητας αυτά, αλλά θα μπορούσαμε ενδεχομένως να εκδώσουμε κατευθυντήρες γραμμές. Σε ορισμένες πόλεις ε, η εισαγωγή νέων τεχνολογιών έχει προχωρήσει πάρα πολύ και ε, ξεχνάνε, ξεχνάμε ε, ότι η επιστροφή σε κάποιες παλιές τεχνολογίες ε, ίσως θα αποτελούσε λύση. Ε, δεν ενισχύουν τόσο πολύ τα αυτοκίνητα σπορ. Γιατί ο αριθμός τους είναι πολύ μικρός. και πάση περιπτώσει αυτοκίνητα, σπόρα αυτοκίνητα μέσα στο κέντρο της πόλης έτσι κι αλλιώς κυκλοφορούν με την ίδια ταχύτητα, κινούνται με την ίδια ταχύτητα με όλα τα υπόλοιπα οχήματα. Οπότε τις ε, ικανότητες, τις δυνατότητες τους χρησιμοποιούν εκτός πόλης πιο πολύ. Ε, συνεπώς ενδεχομένως ε, δεν ενοχλούν τόσο πολύ περισσότερο από ό,τι άλλα οχήματα στις πόλεις. βέβαια, η, η χωμόνωση των δρόμων με παραπετάσματα ε, είναι μια λύση, δεν είναι η βέλτιστη λύση. Προστατεύει αυτούς που κατοικούν μέχρι τον πέμπτο όροφο δίπλα στον αυτοκινητόδρομο. Βέβαια αυτοί που κατοικούν πιο ψηλά ε, δεν προστατεύονται διότι ο θόρυβος περνάει από πάνω από τα παραπετάσματα Ίσως θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε δέντρα ή πρασινάδα, φράχτες, φυσικούς φράχτες, για να κάνουμε λίγο πιο πράσινες και τις πόλεις μας, ε, ε, να, αντί για παραπετάσματα εννοώ, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε ισχυρές ε, ποικιλίε φυτών για φυσική προστασία. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε. Καλή ιδέα τα τρόλεϊ με τα καλώδια και τα λοιπά. Πράγματι είναι και πιο ήσυχα τα ηλεκτροκίνητα οχήματα σχέση με τα υπόλοιπα. Δεν βλέπω κάποιον να ζητάει το λόγο. Α! Κι όμως, ο κ. Ντεμέσμακερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω Ολλανδικά. Μία σκέψη, ε, γιατί είδα αυτό το οποίο είπατε για την αεροπορία και είπατε πως είναι πολιτικά ευαίσθητο ζήτημα. Το επιβεβαιώνω. Ξέρω γιατί πράγμα μιλάω. Εδώ και χρόνια ήμουν μέλος του Φλαμανδικού Κοινοβουλίου εδώ σε αυτή τη χώρα και οι συζητήσεις ε, εξακολουθούν και είναι έντονες για τον Θόρβο. Είχαμε μια κατάσταση ε, που το αεροδρόμιο των Βρυξελών είναι στη Φλάνδρα, ε, αλλά πολύ κοντά στην πρωτεύουσα προφανώς. Και ξέρετε πως η πολιτική ε, του θορύβου είναι κάτι το οποίο καθορίζεται από την περιφέρεια. Κάτι το οποίο κατά κανόνα το βρίσκω καλό, αλλά σε αυτή την περίπτωση είναι παράλογη, παράλογο, γιατί έχουμε την εξή κατάσταση. Στην, στις ε, Βρυξέλλες, στους 19 δήμους είναι πολύ χαμηλές προδιαγραφές του θορύβου Στη Φλάνδρα, εκεί όπου βρίσκεται το αεροδρόμιο, ε, είναι πολύ υψηλότερη η ε, και οι προδιαγραφές είναι πολύ υψηλότερε. Οπότε, τα αεροπλάνα έπρεπε κάποια στιγμή να πάνε σε ένα συγκεκριμένο διάδρομο. Δηλαδή, απογειώνονταν, απέφευγαν τις Βρυξέλλες και έκαναν ένα γύρο. Έτσι. Και ένα μικρό τμήμα του πληθυσμού είχε πολύ μεγαλύτερη επιβάρυνση και δεν μπορούσε πραγματικά να ζήσει. Ξέρω πως είναι ίσως ε, ευσεβής πόθος, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να, ίσως θα μπορούσαμε να το ρυθμίσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί ό,τι γλώσσα και να μιλάνε οι άνθρωποι, ο θόρυβος το ίδιο τους ενοχλεί. Οπότε θα μπορούσε να ρυθμιστεί κάτι τέτοιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο νομίζω. Πράγματι. Η, η, εναρμόνιση είναι καλό. Δεν μπορούσατε να εθετήσετε τις προδιαγραφές των Βρυξελών και στη Φλάνδρα για να λυθεί το πρόβλημα. Ευχαριστώ λοιπόν αυτούς που έκαναν τη μελέτη αυτή και θα δούμε μετά αν θα, αν να το μεταφράσετε και σε άλλες γλώσσες για να υποφεληθεί νομίζω και εκείνη η γνώμη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περνάμε στο επόμενο θέμα εταιρείε χρηματοδοτικής μίσθωσης. Και εδώ πέρα υπάρχει μια μελέτη την οποία θα μας παρουσιάσει ο δόκτωρ Φίλιπ Σέπελμαν από το Ινστιτούτο του Μπατάλ. Έχετε τον ε, λόγο αν είστε έτοιμος. Μπορείτε να ξεκινήσετε. Να ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. η ιδέα του να πουλάμε ε, διάφορα κατά είναι ως ένα βαθμό ξεπερασμένη. Δηλαδή, οι καταναλωτές ενδιαφέρονται για την απόδοση και όχι για την ιδιοκτησία. Οι μεταφορές, ε, φως, ε, η θέση κτλ είναι αυτό το οποίο μετράει. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να έχω στην ιδιοκτησία μου ένα φωτοτυπικό τηλεόραση, hi-fi κτλ. Αρκεί να μπορώ να τα χρησιμοποιώ. Έχουμε λοιπόν τις εταιρείες χρηματοδοτικής ε, μίσθωσης που αποτελούν μια νέα σχέση μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών και βασίζονται σε ένα επιχειρηματικό μοντέλο υπηρεσιών και νέους τρόπους ορισμού των προϊόντων και της ιδιοκτησίας και της ευθύνης. Οι νέες αυτές δομές μπορεί να οδηγήσουν σε ένα σχεδιασμό προϊόντων πιο αποτελεσματικό για να αυξηθεί η ζωή του προϊόντος και να βελτιωθεί η χρήση και θα βελτιώνεται έτσι και η ανακύκλωση. Γι' αυτό είναι, σημα... αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στην Ευρώπη που θα χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους. Οπότε ο στόχος είναι της εταιρείας αυτής να ανταποκριθεί στις ανάγκες των καταναλωτών, όχι να πουλάει προϊόντα. και θα έχουμε και καινοτόμα προϊόντα αλλά και πελάτες οι οποίοι μπορεί να είναι επιχειρήσεις για να οδηγηθούμε σε μια κοινωνία leasing. Αυτό είναι το όραμα και μας ζητήθηκε να εξετάσουμε τους τύπους ε, συστημάτων ε, υπηρεσιών προϊόντων και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα. Βρήκαμε τρεις τύπους συστημάτων υπηρεσιών προϊόντων είναι οι στρατηγικές ε, που βρίσκουμε σε επιχειρήσει. Π.χ. ο καταναλωτής αγοράζει το προϊόν και έχει την ιδιοκτησία του, αλλά μετά υπάρχουν υπηρεσίες μετά την πώληση, π.χ. επισκευές και συμφωνίες επαναγοράς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, αγοράζει κανείς ένα πλυντήριο ή ένα φωτοτυπικό το σε ένα γραφείο Και η εταιρεία που στο πουλάει φροντίζει και τη συντήρηση σε όλο τον κύκλο ζωής του προϊόντος. Μία άλλη στρατηγική είναι στρατηγική προσανατολισμένη προς τον χρήστη. Ο πελάτης αγοράζει την χρήση του προϊόντος και υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι κατανάλωσης και διατηρεί την ιδιοκτησία του προϊόντος. Και πάλι το παράδειγμα εδώ πέρα ε, θα μπορούσε να είναι ένα φωτοτυπικό ή ένα πλυντήριο ε, το οποίο δεν θα πουληθεί στον πελάτη αλλά θα ενοικιαστεί και μετά από λίγο θα παραλάβει ένα καινούριο χωρίς να χρειαστεί να το πληρώσει. Και η τρίτη στρατηγική είναι προσανατολισμένη στα αποτελέσματα. Πουλάμε το αποτέλεσμα του προϊόντος, π.χ. καθάρισμα ή ψήξη ή χαρτί φωτοτυπίας. Οπότε έχει ο παραγωγός την ιδιοκτησία και ο πελάτης έχει μόνο την υπηρεσία. Είχε καθαρά ρούχα ή φωτοαντίγραφα. Και όσο πιο πολύ πάμε προς τις υπηρεσίες, ε, τόσο ε, θετικότερα κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά αποτελέσματα έχουμε. Τα χρόνια που μας πέρασαν, ε, τα επιχειρηματικά αυτά μοντέλα εφαρμόστηκαν στην πράξη και έχουν εδρεωθεί σε κάποια τμήματα της αγοράς και δραστηριότητες business to business. Κάποιες ε, περιπτώσεις ε, αποκαλύπτουν πως συστήματα τέτοιων υπηρεσιών θα μπορούσαν να έχουν ε, κάποια αποτελέσματα και να οδηγηθούμε ε, σε τέτοιες εταιρείες χρηματοδοτικής ε, μίσθωσης και βέβαια αυτό εξαρτάται και από το συνδυασμό των μέσων που έχουμε επιλέξει, το είδος του προϊόντος και το τμήμα της αγοράς που αφορά δηλαδή εξαρτάται το εάν μιλάμε για συναλλαγές μεταξύ εταιριών ή ε, κάποιο λιανικό προϊόν ή προϊόντα μεταξύ καταναλωτών. Το συμβατικό σύστημα του leasing είναι γνωστό, το ξέρετε οι περισσότεροι και οι δραστηριότητε που επεκτείνονται πέρα από τη συμβατική χρηματοδοτική μίσθωση στοχεύουν ε, σε... που θα στόχευαν στις εταιρείες ε, δεν ε, έχουν ακόμα καταγραφεί επαρκώς, αλλά υπάρχουν κάποια επιτυχία αποτελέσματα. Π.χ. υπάρχουν αρκετά παραδείγματα που αναφέρονται στην μελέτη μας, αλλά τα ευρήματα που αφορούν την ποσοτικοποίηση και την εφαρμογή τέτοιων ε, συστημάτων υπηρεσιών και τα οικονομικά και οικολογικά αποτελέσματα, ειδικά στο μακροοικονομικό επίπεδο, δεν υπάρχουν. Οι επιλεγμένες ε, μελέτες ε, συγκεκριμένων περιπτώσεων που έχουμε κάνει είναι βεβαίως περιπτωσιολογία. Ότι κάποιες δηλαδή τέτοιες δυνατότητες υπάρχουν για να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα χρήση των πόρων, ε, αλλά οι μελέτες δεν υποστηρίζουν πως ε, οποιοδήποτε επιχειρηματικό μοντέλο βασίζεται σε ένα σύστημα υπηρεσίας ε, προϊόντων είναι οικολογικά και οικονομικά επιτυχημένο. Βρήκαμε όμως τρεις τάσεις που υπάρχουν παρά το ότι βεβαίως η ιδέα αυτή είναι καινούργια, η υιοθέτηση φαίνεται πως περιορίζεται σε κάποιους κλάδους. Ε, επιτυχείς τέτοιες ε, περιπτώσεις ε, αφορούν συγκεκριμένα τμήματα της αγοράς, π.χ. χημικό leasing, αυτοκίνητα, καθαρισμός χαλιών, διαχείριση εγγράφων και ενέργεια φαίνεται πως ε, υπάρχει βεβαίως μεγαλύτερη διάδοση στον τομέα παροχής υπηρεσιών σε, ε, από επιχειρήσεις σε επιχειρήσεις και από επιχειρήσεις σε καταναλωτές. Όταν μιλάμε για την αξιολόγηση των ε, θετικών και αρνητικών σημείων βλέπουμε πως οι αμοιβαία υποφελείς καταστάσεις εξαρτώνται από το σύστημα για το οποίο μιλάμε και τον κλάδο από τον τύπο του προϊόντος και η μελέτη λέει πως θα μπορούσαμε να έχουμε θετικά οικονομικά και περιβαλλοντικά αποτελέσματα στη μικροκλίμακα, αλλά στην, στο μακροοικονομικό επίπεδο, π.χ. στο ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν φαίνεται κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή. θα μπορούσε να υπάρχει μια σχέση μεταξύ της επιτυχίας αυτών συστημάτων και βελτίωσης ε, για την περιβαλλοντική κατάσταση, αλλά υπάρχουν και άλλες δυνάμεις στην αγορά που εμποδίζουν τέτοια συστήματα και μέσα πολιτικής για να υποστηριχθούν ε, αυτές οι εταιρείε πρέπει να αντιμετωπίσουν αυτά τα ζητήματα εάν είναι να οδηγηθούμε σε καταστάσεις αμοιβαία υποφελής. λοιπόν τα αποτελέσματα καταγράφονται όπως είπα στο μικρό επίπεδο και οπωσδήποτε χρειάζεται ε, περισσότερη έρευνα στο μάκρο επίπεδο για να κάνουμε καλύτερες συστάσεις για τη χάραξη πολιτικής. Παρ' όλα αυτά, μπορούμε να πούμε πως ε, η φύση αυτών των εταιριών και για να είναι μηδέα υποφελής ε, εξαρτάται από τον τύπο της δραστηριότητας και μπορούμε να συστήσουμε κάποια μέσα πολιτικής που θα δημιουργούσαν ένα θετικό πλαίσιο για συγκεκριμένα τέτοια συστήματα υπηρεσίες προϊόντων για να βελτιωθεί η γενικότερη περιβαλλοντική και οικονομική ε, κατάσταση. Το κόστος δε, της πολιτικής αυτής πρέπει να αξιολογηθεί σε ένα δυναμικό πλαίσιο το οποίο θα λαμβάνει υπόψη το αρχικό βεβαίως κόστος ε, εφαρμογής αλλά και την ε, διάχυση που θα έχει και μηχανισμούς ανάδρασης. Και πρέπει βεβαίως να γνωρίζουμε πως ε, μέσα τα οποία θα βασίζονται στην αγορά έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα να οδηγήσουν σε μια μετάβαση σε ένα τέτοιο σύστημα. Τα μέσα τα οποία έχουμε και προτείνουμε δεδομένων των συνδικών και με βάση την αβεβαιότητα που ανέφερα θα δείτε πως είναι αρκετά, τα έχουμε χωρίς μέσα της αγοράς, ρυθμιστικά, μέτρα πληροφόρησης και συμμετοχικά μέσα. Δεν θα μπω τώρα σε λεπτομέρειες. Μπορούμε να συμπεράνουμε πως η χρηματοδοτική μίσθωση έχει τη δυνατότητα να επιφέρει μια επανάσταση ε, σε διάφορους ε, τομείς ε, της κοινωνίας ε, για να οδηγηθεί η Ευρώπη σε μια κοινωνία που θα είναι πιο κοντά στην αποτελεσματική χρήση των πόρων και υπάρχει μεγαλύτερο δυναμικό από τις τεχνολογικές καινοτομίες. Υπάρχουν έτσι κάποια τεχνολογικά ανταγωνιστικά πλέον εκτήματα και θα είναι έτσι η βιομηχανία στην Ευρώπη πιο ανθεκτική και σε εξωτερικούς ε, κινδύνους, ε, σοκ τιμών κτλ. Βέβαια, υπάρχει ο κίνδυνος αποτυχίας εάν προωθήσουμε τα λανθασμένα μοντέλα και θα οδηγηθούμε σε αύξηση της κατανάλωσης ε, ενέργειας και πρώτων υλών. Όλα αυτά λοιπόν απαιτούν μια νέα προσέγγιση στην ανάπτυξη έρευνας και τεχνολογίας, στην αξιολόγηση της τεχνολογίας και στην διακυβέρνηση. Και πρέπει βεβαίω να βεβαιώσουμε εδώ πέρα την έρευνα και την ανάπτυξη. Παρά τι αβεβαιότητε αυτές, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορούσε να κάνει κάποια πρώτα βήματα προς την κατεύθυνση των εταιριών χρηματοδοτικής μίσθωση. Παραδείγματο χάρη, μέσω της εισαγωγή μιας εταιρική σχέσης καινοτομία. Έχουμε τα απαραίτητα μέσα και το θέμα είναι απλά να τα χρησιμοποιήσουμε και να επιφέρουμε κάποια αλλαγή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε, δόκτωρα Σέπελμαν. Δεν έχει ζητήσει κανείς το λόγο. Ε, θεωρώ πως ήταν πάρα πολύ επιτυχημένη η εργασία αυτή. Είναι λυπηρό το ότι αυτοί οι οποίοι ζήτησαν αυτή τη δουλειά δεν βρίσκονται εδώ πέρα σήμερα. Και δυστυχώς έχουν άλλες ανελημμένε υποχρεώσει. Παρόλα αυτά είναι θετικό το ότι ήρθατε εδώ πέρα και μας τα παρουσιάσετε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας ευχαριστώ για την παρουσίαση που κάνετε στου δύο συναδέλφους που είναι ακόμα στην αίθουσα εδώ πέρα μαζί μου. Ε, δεν πρέπει να την πληρώνουν αυτοί που είναι εδώ πέρα, οι απόντε στένε. Σα ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ. Τελειώσαμε αυτό το θέμα στην ημερήσια διάταξη. Η επόμενη συνεδρίαση είναι στι 26 Μαρτίου. Ελία τη συνεδρίαση. Καλώ.